εκπροσώπου για τις εκλογές στη Μιανμάρ. Δίνω το λόγο εξ ονόματος ε, της Αντιπρόεδρου της Επιτροπής, τον Νίκολα Σμιτ, ο οποίος αντικαθιστά την ύπατη εκπρόσωπο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για την παρουσία σας σήμερα το απόγευμα στο Στρασβούργο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στις 8 Νοεμβρίου έγιναν οι ιστορικές εκλογές της Μιανμάρ με συμμετοχή 91 κομμάτων και άνω των 6.000 υποψηφίων. Ο κόσμος ψήφισε υπέρ της αλλαγής και εξέφρασε τη βούλησή του να ζήσει σε μια νέα ελεύθερη δημοκρατική Μιανμάρ. Έδωσαν ξεκάθαρη εντολή στην ΑΕΝ Σαν Σου Κίνγκ, που, οποία ε, της οποίας το κόμμα έχει την πλειοψηφία και στα δύο τμήματα του Κοινοβουλίου της Μιανμάρ, της Βουλής της Μιανμάρ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη δημοκρατική ε, μετάβαση στη Μιανμάρ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο υπ' αυτή την έννοια. Στις 16 Νοεμβρίου η ύπατη εκπρόσωπος τηλεφώνησε στην Aung San Suu Kyi προσωπικά για να τη συγχαρεί για την εκλογική της νίκη και τόνισε πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος των 150 ανεξάρτων παρατηρητών με επικεφαλή στον Αντιπρόεδρο Αλεξάνδρ Λάμστροφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, πόσο σημαντικός ήταν ο ρόλος για τη διενέργεια ειρηνικών και αντικειμενικών εκλογών. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω το μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικότερα για τη συμβολή του στη δημοκρατική αυτή διαδικασία. Ωστόσο, η Ροχινγκίγε και η κατάστασή τους και άλλων, αυτών και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων παραμένουν ε, ζητήματα ανησυχίας. Ε, δεν μπορούσαν να είναι υποψήφιοι ούτε να ψηφίσουν. Μάλλον τα περισσότερα κόμματα ε, υπέκυψαν στις πιέσεις που άσκησαν οι βουδιστές μοναχοί. Στη δήλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρεται ότι οι περαιτέρω συνταγματικές μεταρρυθμίσεις παραμένουν απαραίτητες για απολύτως δίκαιες εκλογές στο μέλλον. Η Aung San Suu Kyi είναι επικεφαλής του μεγαλύτερου κόμματος το Κοινοβούλιο της Μιανμάρα, αλλά βάσει του συντάγματος δεν μπορεί να αναλάβει το αξίωμα της Προέδρου. Ο στρατός θα συνεχίσει να έχει το 25% των εδρών στο Κοινοβούλιο και Τρεις βασικοί υπουργοί θα είναι από το στρατό ανεξαρτήτως του ποια κόμματα σχηματίσουν την κυβέρνηση τελικά. Πρέπει όλοι οι πολιτικοί παράγοντες να ε, εγκαινιάσουν το διάλογο με πνεύμα συμφιλίωσης για να γίνει σωστά η μετάβαση στη δημοκρατία. Παρά τις προκλήσεις αυτές, οι εκλογές ήταν ένα σημείο καμπής. Ήταν τεράστια ευκαιρία να ενισχυθεί η δημοκρατία στη Μιανμάρ. Και στα μέσα Φεβρουαρίου 2016 θα εκλεγεί ο νέος πρόεδρος και θα σχηματιστεί νέα κυβέρνηση μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2016. Παρόλο που η Αούγκ Σαν Kyi δεν έχει ακόμα κάνει προγραμματικές δηλώσεις για τη νέα κυβέρνηση, τα ανθρώπινα δικαιώματα, το κράτος δικαίου και η οικονομική ανάπτυξη θα είναι σίγουρα μέσα στις προτεραιότητές της. Η Μιανμάρ μπορεί να βασίζεται στη δική μας στήριξη. Παραμένουν ζητήματα που μας ανησυχούν και θα συνεχίσουμε επικοδομητικό διάλογο με τη χώρα αυτή. Ε, για παράδειγμα, για το ότι η μειονότητα ροχική για δεν έχει υπηκότητα, ενώ ανησυχούμε και για τη ριζοσπαστικοποίηση των βουδιστών μοναχών και ε, ανησυχούμε για το ότι νομοθετικά έχουν υπάρξει προβλέψεις νομοθετικές για τη φυλή, για τη ράτσα, για τη θρησκεία, για τις θρησκευτικές επεπιθήσεις που δεν συνάδουν με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Μιανμάρ στο επίπεδο αυτό. Το εμπάργκο για τα όπλα αναστάλθηκε το 12 και καταργήθηκε το 2013. Έχουμε το Everything But Arms. Έχουμε εμπορικές προτιμήσεις, ε, συμφωνίες για όλα εκτός από τα όπλα. Αυτά θεσμοθετήθηκαν και θεσπίστηκαν πάλι το 2013. Η Task Force πήγε τον Νοέμβριο του 2013. Η Μίανμαρ ε, επιτάχυνε τη συνεργασία με εμά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έκτοτε. Υπήρχαν δύο γύροι για τα ανθρώπινα δικαιώματα με επικεφαλή του αρμοδίους από πλευράς Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2014 μέχρι σήμερα. Η Μιανμάρ είναι ε, μια χώρα που βρίσκεται ψηλά στι προτεραιότητές μα σε θέματα δημοκρατία και θα ε, ε, παρακολουθούμε εκ το τη συμφωνία που έχουμε με τη χώρα αυτή και που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει μια ευρεία συμφωνία και χειρίας ε, που υπογράφτηκε τον Οκτώβριο του 2015. Με άλλους δωρητές η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί ένα ταμείο για να ενθαρρύνει περισσότερο τη διαδικασία αυτή. Και διαπραγματευόμαστε μια ε, συμφωνία για την προστασία των επενδύσεων και ε, ε, είμαστε μέλος της πρωτοβουλίας για τα εργασιακά δικαιώματα μαζί με άλλους δωρητές ορίζουμε τη στρατηγική μας και θέλουμε να στηρίξουμε τη Μιανμάρ σε αυτή τη δημοκρατική μεταβατική διαδικασία. Και όλα αυτά υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων στα συμπεράσματά του τον Ιούλιο του 2015 μεταξύ άλλων. Προτεραιότητες μας είναι η ειρήνη, το εμπόριο, η δημοκρατία, η ανάπτυξη και η, η παρουσία της Μιανμάρ στη διεθνή κοινότητα με επιτυχία. Με το πολιετές ενδεικτικό πρόγραμμα δράσης της Μιανμάρ 2014-2020 ε, το προπολογισμό θα είναι 688 εκατομμύρια που θα δοθούν για μέτρα οικοδόμησης της ειρήνης, για το κράτος δικαίου, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τις ε, οικονομικές και αναπτυξιακές μεταρρυθμίσεις. Δίνουμε ανθρωπιστική βοήθεια στα πιο ευπαθή τμήματα του πληθυσμού και κυρίως ε, στους εκτοπισμένους μεταξύ άλλων οι δεσμεύσεις μας εκτείνονται σε ένα μεγάλο φάσμα και αυτό δείχνουν τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τον εκδημοκρατισμό της χώρας αυτής. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το παν ώστε η μετάβαση στη δημοκρατία ε, της Μιανμάρ να φτάσει σε, ε, στο τέλος της με επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε ε, κύριε Υπουργέ. Τώρα περνάμε τις ομάδες. Ο πρώτος ομιλητής είναι ο κύριος Αντάκουσον ε, από το ΕΛΚ. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε στην κατάσταση, να παρακολουθήσουμε δηλαδή την εκλογική διαδικασία στη Βυρμανία. Τα αποτελέσματα είναι θετικά ως, ε, δηλαδή ως προς την διενέργεια των ε, εκλογών και την καταμέτρηση. Είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα, δεν υπήρξε νοθεία και η συμμετοχή ήταν της τάξης του 80%. Η Αν εκεί και το κόμμα της, το κόμμα έλαβε την πλειοψηφία και θα πρέπει να δημιουργηθεί νέα κυβέρνηση. Θα πρέπει λοιπόν οι εκλογές στη Μιανμάρ να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο. Έχει επιτευχθεί πολιτική πρόοδος, όμως η χώρα αυτή δεν είναι πραγματική δημοκρατία. Το Σύνταγμα εμπεριέχει διατάξεις που προβλέπουν ότι οι στρατιωτικοί μπορούν να κατέχουν το 1 τέταρτο των ευρών του Κοινοβουλίου και η Aung δεν μπορεί να ε, οριστεί πρόεδρος γιατί κατέχει και τη Βρετανική υπηκότητα. Υπάρχουν μεγάλα προβλήματα με την μειονότητα των Ροχίνια, οι οποίοι είναι μία μουσουλμανική μειονότητα. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Θα πρέπει να υπάρξει εθνική συμφιλίωση για να μπορεί να κινηθεί η Μιανμάρ προς τη σταθερότητα. Από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες η κυρία Κόμες έχει το λόγο για δύο λεπτά. Επειδή συμμετείχα στην Επιτροπή Παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να ευχαριστήσω γιατί μπόρεσα να παρευρεθώ στις πιο ανοιχτές εκλογές μετά από 60 χρόνια σειράξεων και 50 χρόνια δικτατορίας. Και αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι το Σύνταγμα το οποίο ε, επιβλήθηκε από την στρατιωτική χούντα το 2008 επιβάλλει ώστε το 1 τέταρτο των εδρών να κατέχουν οι ίδιοι στρατιωτικοί χωρίς να υποβάλουν υποψηφίους για να μην μιλήσουμε για εκατομμύρια πολιτών εθνοτικών μειονοτήτων που δεν έχουν καν εγγραφή στα Μητρώα. Παρόλα αυτά έχει ε, επιτελεστεί πρόοδος, αν μη τι άλλο λόγω της ε, κατήσχησης του κόμματος της Ανσανσουκή και της ε, κατάρρευσης του κόμματος των στρατιωτικών. Ελπίζω να υπάρξει πραγματικά εθνική συμφιλίωση και ειρήνη. Δεν είναι κάτι το εύκολο σε ένα στρατιωτικό ε, καθεστώς, μέχρι τώρα στρατιωτικό καθεστώς, όπου οι στρατιωτικοί ε, κατέχουν θέσεις κλειδί και όπου οι Ροχίνγκια δεν μπορούν ούτε να ψηφίσουν ούτε να υποβάλουν υποψηφιότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι ξενοφοβικοί βουδιστές ε, έχουν αποτρέψει αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει πολύς ρατσισμός και διακρίσεις από τους μοναχούς βουδιστές και γι' αυτό θα πρέπει να επιβάλλουμε την τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε την ε, υπερίσχυση της δημοκρατίας και να υποστηρίξουμε και το NLD και την κοινωνία των πολιτών, έτσι ώστε να αλλάξει και το Σύνταγμα. Από τους Ευρωπαίους Μεταρρυθμιστές και Συντηρητικούς, ο κύριος Τάνοκ. Η νίκη του LND είναι ένα ιστορικό ορόσημο, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το, ε, τη δράση του USDP. Ξέρετε τι συνέβη το 1990. Η δημοκρατική μετάβαση τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολη και θα πρέπει να υποστηρίξουμε την τρέχουσα κατάσταση θα πρέπει να μας απασχολήσει και το θέμα των στρατιωτικών που κατέχουν το 25% των εδρών στο Σύνταγμα και το κόμμα της Ανσανξουκή στην ουσία υποβαθμίζεται γιατί η ίδια δεν μπορεί να αναλάβει ε, την Προεδρία επειδή κατέχει και τη Βρετανική υπηκότητα. Επίσης, οι μουσουλμάνοι Ροχίνγκια, ένα περίπου εκατομμύριο, δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε εκλογές και δεν έχουν κάνει ηθαγένεια. Η Ανσάν δεν είπε και πολλά για το θέμα και το NLD, το κόμμα της, δεν θέλει να, να βελτιώσει την κατάσταση των Ροχίνγκια μέσα στα πλαίσια του εκδημοκρατισμού Ανμάρ. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά νομίζω ότι το Μιανμάρ θα φτάσει σε μια πλουραλιστική δημοκρατία. Αυτή η μετάβαση στη δημοκρατία είναι ευπρόσδεκτη μέσα στα πλαίσια της δημοκρατικής αξιοπιστίας της Ασίας. Από τους φιλελευθέρους, ο Αντιπρόεδρος Λάμστορφ έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε πρωτεύουσα του Συμβουλίου σας, ευχαριστώ για τις ε, γενικέ σα κουβέντε και φαντάζομαι ότι αυτό είναι έπινο για όλη την ε, αποστολή. Μέχρι την ε, τελική έκθεση έχω εντολή, γι' αυτό λοιπόν θα χρησιμοποιήσω αυτή την αρχή του κεντρικού παρτρίτη. Ήταν πραγματικά ιστορικές οι εκλογές και όποιο έχει πολιτική διέστηση αντελήφθησε τι ελπίδα ε, γεννήθηκε από τις εκλογές αυτές στη χώρα. Και ήταν καλό που μπόρεσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση από πριν αλλά και με την ε, αποστολή παρατηρήσει να συμβάλλει. Και χαίρομαι για δύο πράγματα. Καταρχάς, ε, ότι δεν υπήρχε σχεδόν καθόλου βία στις εκλογές, ούτε πριν ούτε μετά. Κατά δεύτερον, πολλά από τα προβλήματα τα οποία υπολογίζαμε ότι θα παρουσιάζονταν την ημέρα των εκλογών δεν παρουσιάστηκαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα, η μεγαλύτερη ανησυχία είναι ε, το ότι δεν υπήρξε πρόβλημα με τις καταλόγους των ε, ψηφοφόρων και το αποτέλεσμα αυτό ο Τσάλς Τάνακ μίλησε για μια περίεργη συνταγματική κατάσταση, αλλά αυτό το συζητήσαμε και προκαταρτικά. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτό φέρνει σε μια πολύ ευαίσθητη μεταβατική φάση τη χώρα και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να παραμείνει δεσμευμένη στη χώρα αυτή και να βοηθάει τη χώρα αυτή και στο μέλλον. Και να πω ανοιχτά το εξή. Ασκείται κριτική για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό ισχύει και εδώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αντιπροσωπεία, η κυρία Σαρτζεντίνη, η οποία είναι μόνιμη εισηγήτρια και θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη χώρα. Ήταν εξαιρετική συνεργασία της με την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τα Μέσα Εξωτερικής Πολιτικής και κυρίως με την Αποστολή. Ήταν πραγματικά εξαιρετική η συνεργασία με τον Λαν Κομπιά. Ένα πολύ καλό παράδειγμα για την καλή λοιπόν συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα συνεχίσει τον καλό δρόμο η χώρα με την δέσμευση και των Ευρωπαίων. Ευχαριστώ. Τώρα για τους πράσινους λέει ο Πρόεδρος. Το λόγο έχει η κυρία Σαρτζεντίνη για ένα μισό λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η κριτική για την προετοιμασία των ε, εκλογών έγινε από τους συναδέλφους Όντω πάρα πολλά άτομα δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν και συμφωνώ με την ανάλυση του συναδέλφου Τάνοκ για το κατά πόσον η κυρία Σαν Σουκί θα δώσει όσα χρειάζεται για τις μειονότητες. Αλλά παρά την κριτική αυτή, βλέπα, είδαμε ότι οι εκλογές διοργανώθηκαν με εξαιρετικό τρόπο. Και κυρίως οι νέες γυναίκες οι οποίες ήταν στα εκλογικά κέντρα πρέπει να πω ότι αξίζουν ιδιαίτερου ε, επένου, αλλά και κάθε μέρα διοργανώνουν εκλογέ. Και βλέπαμε, είδαμε επίση ότι ε, αποδέχθηκε ο στρατό την ε, νίκη του NLD μετά τις εκλογές και αυτό αποτελεί μια πολύ καλή αρχή για μια τέτοια νέα δημοκρατία αλλά δεν έχουμε ακόμα φτάσει στο στόχο αυτό εδώ και 25 χρόνια προσπαθούν οι στρατιωτικοί να φέρουν τη χώρα στην φάση αυτή όπου μπορούμε πλέον να μιλάμε για δημοκρατία και αυτό είναι μια κατάσταση στην οποία μπορούμε να δραματίσουμε ένα ρόλο και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και το Μιανμάρ συμφωνήσαμε ότι αποτελεί μία από τι χώρε ε, στι οποίε θέλουμε να βοηθήσουμε την κοινοβουλευτική δημοκρατία και είναι δικό μου καθήκον αυτό με την δική σα βοήθεια. Είναι μεγάλο αυτό ω όγκο δουλειά. Πρόκειται για μια βουλή όπου κάθονται όχι ένα αλλά αλφαβητικά οι βουλευτές. Καταλαβαίνετε, έχουν πολλά ακόμα να γίνουν. Ο Μπετίνη. Ευχαριστώ. Και εγώ συμμετείχα στην αποστολή παρατηρητών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που παρακολούθησε τις εκλογές στη Βυρμανία υπό την αιγίδα της εξαιρετικής συναδέλφου Γκόμες το κόμμα της Aung San Suu ε, κατάφερε να ε, κερδίσει με τρία βασικά Υπουργεία των Εσωτερικών, Άμυνας και Εξωτερικών. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντιμετωπίστηκαν ε, οι δυσκολίες και παρόλα αυτά οι εκλογές διαξήχθηκαν κανονικά με τη συμμετοχή ενός θαραλέου λαού ο οποίος άδραξε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Όμως παρά το γεγονός ότι γίνεται μετάβαση, η μετάβαση αυτή είναι επώδυνη και θα πρέπει να είμαστε Είμαστε πολύ προσεκτικοί μέχρι την τελική ανακοίνωση των ε, αποτελεσμάτων. Θα φτάσουμε λοιπόν, σε, θα περάσουμε σε μία διακυβέρνηση όπου δεν θα συμμετέχουν στρατιωτικοί. Και μην ξεχνάμε και τον ηρωισμό της Σαν Σανξουκή, η οποία ε, υπέστη βασανιστήρια όπως πολλοί δημοκράτες. Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το παλαιό καθεστώς δεν θέλει να αφήσει την εξουσία. Η Βυρμανία θα υποστηριχθεί. Εγώ βρήκα στους καταβλισμούς πολλούς απάτριδες στα σύνορα με την Ταϊλάνδη όπου ε, ζούσαν πραγματικά σε αχυροκαλύβες χτισμένες πάνω στη λάσπη. Όμως οι Βυρμανοί περιμένουν πολλά από μας και δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε. Γκέρλινγκ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εκλογικός θρίαμβος της Αουν Σαν είναι λόγος πραγματικά για ε, εορτασμό. 77% πήρε στις εκλογές και σίγουρα αυτό θα σημαίνει την αλλαγή στη Μιανμάρ. Οι προκλήσεις είναι σημαντικές. Οι εθνοτικές μειονότητες έχουν πολλά προβλήματα. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουν. Και παρόλο που ο στρατός και οι αντίπαλοι συμφώνησαν να σεβαστούν το αποτέλεσμα των εκλογών, η πραγματική πρόκληση είναι ποια θέση τελικά θα καταλάβουν αυτές οι δυνάμεις στο, στην επόμενη μέρα για ένα καλύτερο μέλλον. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμβάλλει. Να αξιοποιήσουμε αυτή τη διαδικασία όχι μόνο για να ενισχύσουμε την πορεία της Μιανμάρ στη δημοκρατία αλλά και για την ενθάρρυνση των σχέσεών της με τις υπόλοιπες χώρες που είναι μέλη της Ένωσης χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας. Ως μέλος της αντιπροσωπείας ΑΣΕΑΝ είχα το προνόμιο να επισκεφθώ την Aung San Suu Kyi στο σπίτι της πριν από κάποια χρόνια. Ήταν από τις πιο σημαντικές στιγμές στην πολιτική μου σταδιοδρομία. Την ε, συγχαίρω για την πραγματικά μεγάλη εκλογική της επιτυχία. Ο κύριος Μποστινάρου, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη... τη συμπαράστασή μου στις οικογένειες των θυμάτων των εργατών που έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα. Βεβαίως οι εκλογές αυτές ε, είναι πολύ σημαντικές και χαιρόμαστε διότι η εκλογική διαδικασία διενεργήθηκε ομαλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να εκφράσει τη βούλησή του και ο κόσμος πραγματικά εξέφρασε τη στήριξή του στη δημοκρατική διαδικασία. Τα επίσημα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο λαός της Μιανμάρ στήριξε ε, ένα σύμβολο ειρηνικής διεκδίκησης της δημοκρατίας που είναι η Aung Σαν Suu που έχει κερδίσει το βραβείο Σακχάροφ αλλά και το Νόμπελ Ειρήνης. Οι εκλογές αυτές είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης. Αυτό μόνο όμως, γιατί η μεταβατική δημοκρατική διαδικασία θα είναι μακρά το 20%, το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου θα πάνε στο στρατό. Δεν μπορεί ο Αουνξάν να καταλάβει τη θέση του Προέδρου παρόλο που έχει κερδίσει τις εκλογές και θα πρέπει υπουργικά αξιώματα να καταλάβει ο στρατός επίσης. Το σημαντικό είναι να ξεκινήσει μια διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης με ενθαρρύνει το γεγονός ότι ο στρατός αναγνωρίζει το αποτέλεσμα. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για την έλευση των μεταρρυθμίσεων. Να είμαστε ενωμένοι όλοι ως Ευρώπη δίπλα ε, στη χώρα αυτή. Ο κύριος Τζιλ, να... Η κυρία Τζιλ για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σημαντικό σημείο καμπής ε, ήταν οι εκλογές αυτές στη Μιενμάρ. Και έχουμε και τις ε, αποστολές των ε, ανεξαρτήτων παρατηρητών των εκλογών από πλευράς Ηνωμένων Εθνών, τις οποίες διάβασα προσεκτικά. Συγχαίρω την Αουν Σαν Σουκί για την νίκη της. Παρ' όλα αυτά οι ανησυχίε παραμένουν. Οι Ροχινγκίγια δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν. Η νομοθεσία με βάση τη φυλή ή τη θρησκεία σε καμία περίπτωση δεν συνάδει με τη διαδικασία εθνικής συμφιλίωσης. Το περασμένο Σάββατο μάθαμε ότι άνω από 100 άτομα πέθαναν σε μια κατολίσθηση ε, κοντά σε κάποιο ορυχείο, νεφρίτη. Και Ε, ε, σειράξεις, συγκρούσεις όπως αυτή στο Ανατολικό Κονγκό μας έχουν διδάξει ότι η ειρηνή δεν είναι ε, εφικτή πριν κοπεί αυτός ο γόρδιος δεσμός μεταξύ στρατιωτικού σκέλους και εμπορικής οικονομικής δραστηριότητας από την άλλη. Πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να στηρίξει τη νέα πολιτική ηγεσία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα και να ενταχθεί στη δυναμική της ΑΣΕΑΝ, των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Βλέπουμε χώρες πολύ σημαντικές, όπως η Μαλαισία, να πιστοχωρούν σε ό,τι έχει να κάνει με τα ανθρώπινα δικαιώματα τελευταία και αυτό είναι πολύ δυστυχές. Ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν υπάρχει κάποιος από την Επιτροπή εδώ ή κάποιον, κάποιος τέλεχος της είπα της εκπροσώπου, να μας βοηθήσει και να μας ενημερώσει για το πώς γίνεται ο συντονισμός όλων των πολιτικών έτσι ώστε ε, το εμπόριο και οι επενδύσεις να ενισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να μην τα υπονομεύουν. Και οι σχετικές συμβάσεις και συμφωνίες που έχουμε σε αυτό το πλαίσιο εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία Eye, ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σχολιάσω και να επενέσουν την Μιανμάρ για τη διεξαγωγή εκλογών με ιστορική σημασία. Οι πολίτες της Μιανμάρ ε, ψήφισαν και έδειξαν ποια ήταν η θέλησή τους και αυτό μεταφράστηκε σε δημοκρατία. Το βασικό μου ερώτημα είναι τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Η διαδικασία προσέγγισε τη χώρα στη δημοκρατία. Αλλά πολλά ακόμα απομένουν να γίνουν. Θέλω να πιστέψω ότι το NLD θα, σταματήσει, θα ξεκινήσει τη διαδικασία μεταρρύθμισης στο Μιανμάρ. Η εθνική συμφιλίωση και η συμπερίληψη όλων είναι θέματα τα οποία όμως θα πρέπει να είναι στην κορυφή των προτεραιοτήτων και αυτό θα αποτελέσει βασική πρόκληση για την κυρία Σανσου Κι. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μεγάλη εμπειρία με τέτοιες διαδικασίες ε, μεταβατικές και όσο εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε σε θέση και διατεθειμένοι να συνδράμουμε στην, τους φίλους μας στη Μιαμάρ. Θα ήθελα να είμαστε έτοιμοι για να παρέχουμε αρρωγή προς τη χώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ο κύριος Νοτσιμαγιάς. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο λαός της Μιανμάρ στις εκλογές της 8 η Νοεμβρίου αποφάσισε να θέσει τέλος στην κυριαρχία των στρατιωτικών και της Χούντας που κυριαρχούσαν στη χώρα τα τελευταία 25 χρόνια. Εκατομμύρια πολίτες συμμετείχαν μαζικά στις γενικές εκλογές και έδωσαν τη νίκη στην Αούγκ Σαν Σουκί, τη βραβευμένη με Νόμπελ ειρήνης πολιτικό που έχει υποστεί διώξεις από τη Χούντα της Μιαμάρ. Όμως η νέα δημοκρατική κυβέρνηση έχει μπροστά της σημαντικές προκλήσεις. Πρώτα απ' όλα οι στρατιωτικοί πρέπει να πάψουν να κατέχουν το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου. Δεύτερον πρέπει να καταργηθεί η λογοκρισία ταυτόχρονα πρέπει να εξαλειφθεί η καταναγκαστική εργασία ο ρατσισμός και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να σταθεί στο πλευρό της νέας δημοκρατικής κυβέρνησης της μιανμάρ η οποία όμως κυβέρνηση πρέπει επιπροσθέτως να διασφαλίσει και την προστασία των εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν στη χώρα όπως η ροχίνγκια σε βάρος των οποίων συνεχίζονται οι διακρίσεις και η καταπίεση από τους βουδιστές όπως έχω καταγγείλει επανειλημμένα στην αίθουσα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, Ο κύριος Καστάλντο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι εκλογές αυτές στη Μιανμάρ μας μιλούν για μια σοβαρή μετάβαση προς τη δημοκρατία και θα ήθελα να ευχαριστήσω ευχαριστήσω τους συναδέλφους που εκπροσώπησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε μια ιστορική στιγμή. Τώρα, ενώπιον της κυβέρνησης του Μιανμάρ υπάρχουν σοβαρές προκλήσεις. Θα πρέπει να μειωθεί η επιρροή των στρατιωτικών που κατέχουν το 25% των εδρών του Κοινοβουλίου. Ε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σε αυτή τη χώρα ε, μόνο το 1,8% δαπανάται στην υγεία και το 0,8% για την εκπαίδευση. Η ευημερία έχει μεγάλη σημασία καθώς και η καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις κατά τον Ροχίνγκια η Αν μιλάει για το φόβο που είναι και η μόνη φυλακή. Ελπίζουμε να μην φυλακιστεί έναντι των αλλαγών το Μιανμάρ. Ελπίζουμε να ανταποκριθεί στις αλλαγές. Ο κ. Πόλτσακ έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Και πρέπει να ομολογήσω ότι σήμερα το πρωί όταν ε, ενημερωθήκαμε για τα εκλογικά αποτελέσματα. Ήταν πραγματικά μια θαυμάσια στιγμή όπου μπορέσαμε να θαυμάσουμε την πρόοδο της Μιανμάρ τα τελευταία χρόνια. Κατανοώ τις επικριτικές ε, παρατηρήσεις που έγιναν σε σχέση με τη συμμετοχή κάποιων θετικών ομάδων, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε τη διαδικασία που ξεκίνησε στη Μιανμάρ. Και επίσης θα πρέπει να υποστηρίξουμε και την ε, νικητρία σου Σουκί που πλέπει πλέον αναλάβει την ε, πρόοδο. Έχει την ευθύνη αυτή. Θα πρέπει λοιπόν να καταβάλουμε και να υποστηρίξουμε τις προσπάθειες εκδημοκρατισμού γιατί βλέπουμε το θάρρος που έχει επιδείξει ο κόσμος εκεί. Βλέπουμε τα χαρούμενα πρόσωπά τους. Θα πρέπει να τους υποστηρίξουμε λοιπόν για την κοινό μας συμφέρον που το επιτάσσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Και έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται η συζήτηση, λέει ο Πρόεδρος. Και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι οι Ισπανικές Αρχές μας ενημέρωσαν, ενημέρωσαν μάλλον τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι ο κ. Καβιεμπενιτο Ζουλιάκα εξελέγει ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και